Την ημερήσια διάταξη θα τη βρείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.